Δεν έχουμε πολλές. Έκθεση του κυρίου Μωράιες για την αυτοπομημένη ανταλλαγή στοιχείων για τις άδειες κυκλοφορίες οχημάτων στη Λετωνία. Ονομαστική ψηφοφορία η οποία και άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη, έκθεση Γκρίσμπεκ, τεκμήρο αθότητας και δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη για ποινικέ διαδικασίες. Πρώτα ψηφίζουμε το μπλοκ 1, τοπολογία 52, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπλοκ 2, καταπίπτει. Ψηφίζουμε την πρόταση της Κομισιόν, ε, ανατάσσεως χειρός υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα, ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην έκθεση της κυρίας Φόρντ για τα μέσα ατομικής ε, προστασίας. Ψηφίζουμε το μπλοκ 1, τροπολογία 158, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πλοκ 2 καταπίπτει πρόταση της Επιτροπής Διανατάσεως της Χειρός υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για την ε, πρόταση νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Στήλερ για συσκευές αερίου. Ψηφίζουμε το μπλοκ 1, τροπολογία 203. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου με ονομαστική οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Λόπες Στούρες Βάιτ για εγκαταστάσεις σύρματοσχήνων. Μπλοκ 1, τροπολογία 148 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πρόταση της Επιτροπής υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται και η ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Πέρας και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Τώρα περνάμε στις πρότασεις ε, ψηφίσματος αντίρρηση επί του κατεξοδότης κανονισμού για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Ψηφίζουμε το ψήφισμα καταρχήν των ομάδων με ονομαστική οποία και αρχίζει. Της Γκουε. Πέρας. και απορρίπτεται. Πράγμα στην επόμενη έκθεση που αφορά την αντίρρηση επί της καθεξοδότησης πράξης σε σχέση με τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και παιδικές τροφές. Ε, ο κύριος Τέιλορ θα ήθελε να μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έχετε το λόγο. Η ψηφοφορία αυτή αφορά τα κατά πόσο θέλουμε να προωθήσουμε την επιδημία της παχυσαρκίας ή να προστατέσουμε την υγεία των παιδιών και των μελλοντικών γενεών. Η Επιτροπή πρότεινε να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε 30% περιεκτικότητα σε, σε ζάχαρη των παιδικών τροφών και αυτό είναι απαράδεκτο σε σχέση και με τις συστάσεις του ΠΟΗ γιατί μιλούν για ελεύθερη ζάχαρη κάτω από 10% της ε, συνολικής ενεργειακής πρόσληψης και κάτω από 5% ε, για ε, υπέρ της υγείας των παιδιών. Γι' αυτό θα ήθελα να προβάλλουμε αυτή την πρόταση έτσι ώστε να συμβαδίζει με τις συστάσεις του ΠΟΗ. έτσι ώστε όλα τα παιδιά της Ευρώπης να έχουν ένα υγιέστερο μέλλον. Θα ήθελα να υπερψηφίσετε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Ε, τώρα ο Επίτροπος Χανιέται έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, η έγκρεση της κατεξιοδότηση πράξης αμελήτη ε, δημιουργεί ε, μία συμφωνία με βάση αυτά που είχε ορίσει ο νομοθέτης για τις 20 Ιουλίου 2015. Η κατεξιοδότηση πράξη ορίζει σαφέστερους ε, κανόνες έτσι ώστε οι παρασκευαστές να μπορέσουν να ανταποκριθούν ιδιαίτερα στον τομέα της σήμανσης. Η Επιτροπή δέχεται τη δέσμευση των υπηρεσιών για να έρθουμε σε επαφή με την ΕΦΣΑ μέχρι τα τέλη του 2016 σε σχέση με την περιεκτητή ποσοτικότητα των τροφίμων με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές σε σχέση με τα επίπεδα ε, ζάχαρης. Με βάση του στόχου της ΕΦΣΑ, του Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων, θα μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε την περιεκτικότητα αυτών των παιδικών και άλλων τροφών. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Τώρα αρχίζουμε με τροπολογία 2 με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Το αρχικό κείμενο. Διανατάσεως υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Αρχικό κείμενο. Δεν είσαστε σίγουροι, θέλετε να ελέγξουμε την παράγραφο 3. Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται πράγματι. Παράγραφος 4. Αρχικό κείμενο διανατάσεως υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Όχι, έχουμε την ίδια την ίδια πλειοψηφία. τρία υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ένα Πρώτο τμήμα του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη F σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη G. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και η πρόταση στο σύνολό της, πρόταση ψηφίσματος μονομαστική, η οποία και αρχίζει. Πέρας. Και εγκρίνεται. Η Ειρηνευτική διαδικασία για την Κολομβία. Έχουμε μια κοινή πρόταση ψηφίσματος, είναι και η τελευταία πρόταση. Ψηφίζουμε διανατάσεως το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος περ κατά αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Λίγη διαδικασία ψηφοφοριών. Περνάμε στις αιτιολογήσεις ψήφου.